ασκούν ε, κάποιοι, ε, δεν ναι, ε, υπάρχει ασυμβίβαστο. Περνάμε τώρα σε παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζαμπόσκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να θυμίσω ότι από χθες ξεκίνησε, ε, ετέθησαν ε, νέα ανώτατα σημεία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρί ε, μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα ήταν δυνατόν δεν υπήρχε μια στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για μέτρα τα οποία αφορούν τον κάθε πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα, τους τελευταίους οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν αντικείμενα επικρίσεων. Είμαι πεπισμένη ότι το ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο ε, έχει κάποιο νόημα. Είναι σημαντικό αντί να διεξάγονται ανώφελε συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωνόμαστε σε πρακτικά προβλήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαζίτ Ιλτάλγκο έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, είμαι βαθιά συγκινημένος διότι συνάντησα τους ανθρακορίχους που έκαναν πορεία στη Μαδρίτη και είδα ότι πραγματικά η Ισπανική κυβέρνηση δεν ακούει. Η αιώνια Ισπανία είναι η αξία την οποία προέβαλαν οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, οι αιώνιες αξίες της χώρας μας, της χώρας μας εκπροσωπούνται από τους ανθρακορίχους, από τα ορυχεία, από αυτή την ανάγκη και δυνατότητα αντίστασης, οι οποίοι πριν από 50 χρόνια ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στη δικτατορία του Φράνκο και έτσι έκαναν το αποφασιστικό βήμα για την ελευθερία. Κάθε φορά που γίνεται λόγος για τον Σαλβαδόρ Ντεμαραδαριάγα όλοι γνωρίζουμε, όλοι γνωρίζουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, εξού και υπάρχει κτίριο αφιερωμένο στο όνομά του προς τιμή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στη συνέχεια στον κύριο Κριστιαν Μπιζόη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για την οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίπτωση που έχει στη Ρουμανία. Μία ευφυής πολιτική για τα φάρμακα μας χρειάζεται οπωσδήποτε, μια καλή πολιτική για την εμπορία των νέων προϊόντων, ο καθορισμός των τιμών, η επιστροφή του κόστους των φαρμάκων για πολλούς πολίτες της Ένωσης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Στην Ρουμανία Κάποιες ατυχείς αποφάσεις ελήφθησαν μεταξύ 2009 και Απρίλιο 2011. Υπάρχει ένας κατάλογος των φαρμάκων που καλύπτονται ε, που ισχύει για τέσσερα χρόνια όμως και εξαρτάται από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Όταν αναπτύσσονται καινούργια μόρια, δραστικέ ουσίες, ε, ε, μπορεί τα μέτρα να είναι πολύ αυθαίρετα. Η εμπορία κάποιων φαρμάκων στη Ρουμανία ε, εμποδίστηκε λοιπόν στη Ρουμανία μετά το 2011 παρακαλώ την Κομισιόν να προσέχει πιο πολύ αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα. Κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να εκφράσουμε την μεγάλη μας ε, απογοήτευση λόγω του πραξικοπήματος στην Παραγουάη. Ε, έχασε τη θέση του Προέδρου ο κύριος Φερνάντο Λούγο βάσει μιας διαδικασίας η οποία δεν τηρεί τις δημοκρατικές δεσμεύσεις, δεν δόθηκαν 24 ώρες για να προετοιμαστεί και είχε μόνο δύο ώρες για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Όλα αυτά ήταν παράνομα, αντιθεσμικά, αντισυνταγματικά και τελικά έγινε χειραγώγηση της Δημοκρατικής Βούλησης η οποία βούληση του λαού αποφάσισε να αλλάξει ε, την κατάσταση στην Παραγουάη μετά από 40 χρόνια δεξιάς κυβέρνησης. Θα πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Στην Παραγουάη έγινε κοινοβουλευτικό ε, πραξικόπημα και το οποίο ε, καταδίκασε και η Μερκοσούρ και διάφορα άλλα πολύ σημαντικά διεθνή θεσμικά όργανα γίνεται αυτή τη στιγμή μια πολιτική δίκη εναντίον του Προέδρου της Παραγουάης. Θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να πούμε ότι δεν είναι το πλήγμα εναντίον του Φερνάντο Λούγο, είναι το πλήγμα ενάντια ε, στη, στην δημοκρατική διαδικασία και στην δημοκρατία γενικώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλίδης έχει το λόγο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο θέμα της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τηρεί μια ενωμένη στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την Τουρκία όσον αφορά το πεδίο της εφαρμογής της ελόγω συμφωνίας. Όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου σχετικά με την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Τουρκία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η ευρωπαϊκή επιτροπή και το συμβούλιο αναμένουν η τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία με αμερόληπτο τρόπο εναντί όλων των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής δημοκρατίας. παρεμπιπτόντως γιατί προβλέπεται μια περίοδος χάριτος τριών χρόνων στην τουρκία όσον αφορά την επανεισδοχή υπηκών τρίτων χωρών αυτή η πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών χαλάει τη συνέπεια της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό και μπορεί να βλάψει τις σχέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης με τις άλλες τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το θέμα. Ξέρουμε ποιο δεν θα είναι το θέμα. Θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, κανένας δεν το ξέρει. Όλοι μας εδώ ξέρουμε ότι θέλουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε της Η κρίση τη Ευρωζώνη χρησιμοποιείται για να, για να υπάρξει πλήρη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο μόνο που δεν το καταλαβαίνει αυτό είναι ο Ντέιβιτ κάμερον ή το ανεξάρτητο ε, κόμμα μπορεί να το εξηγήσει όπως το για να το εξηγήσει και τους, στους ψηφοφόρους. Αυτό που θέλουμε ε, για δημοψήφισμα είναι θα πρέπει να μείνουμε ή να φύγουμε και είναι καλύτερα να γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Μπάτιν, ο κύριος Ζεγκεντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για ένα μικρό οικισμό στην Ουγγαρία που λέγεται Όνοντ. Εμείς οι Ούγγροι είμαστε πολύ περήφανοι για το μικρό αυτό οικισμό στο Όμπους Σέμπλιν γιατί πριν από 300 χρόνια έγινε στο Όνοντ μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική συνέλευση και τώρα για πολλά χρόνια έχουμε και ε, ένα, μια πολύ φημισμένη ε, γιορτή εκεί. Το Όνοντ ε, υπετάχθη στους ε, Τούρκους, στους ε, Αψβούργους και στο κομμουνιστικό καθεστώς. Όμως αναφέρομαι σε, κάποιους, σε κάποιες φήμες που λένε ότι δεν συνάδει η γιορτή μας με το κοινοτικό δίκαιο. Μην θυσιάσουμε παρακαλώ το όνοντ στο βωμό του ελευθέρου εμπορίου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το Όνοντε είναι ένας χώρος όπου μικροί έμποροι μπορούν να έρχονται ε, να ανταλλάσσουν τα εμπορεύματά τους, ε, μικροί κτηνοτρόφοι. Τέτοια ε, πανηγύρια θα πρέπει, τέτοιες πανηγύρις θα πρέπει να διατηρηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαπερκόφσκι δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σικέρσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα το τελευταίο σφύριγμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, των εθνικών ομάδων δηλαδή. Ολοκληρώθηκε το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική μαζική εκδήλωση, η πιο μεγάλη αθλητική διοργάνωση που έχουμε οργανώσει ποτέ εμείς στην Πολωνία και είμαστε περήφανοι για την επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της αθλητικής διοργάνωσης. Έχει πνεύσει ένας νέος αέρας στη χώρα μας όχι μόνο στο χώρο των αθλημάτων, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι όλοι όσοι ταξίδεψαν στην Πολωνία και στην Ουκρανία εκτίμησαν ιδιαιτέρως τη διοργάνωση, τη φιλοξενία, το ήρεμο πνεύμα, τη φιλική διάθεση και θέλουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη που μας επιδείξατε και για τη στήριξη που μας προσφέρατε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βοήθειά της η οποία μας επέτρεψε να βελτιώσουμε τις οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές μας οι οποίες χρησιμεύσαν όχι μόνο για την αθλητική διοργάνωση αλλά θα χρησιμεύσουν και στο λαό μας, στους λαούς μας, στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Καστέξ. Κυρία Πρόεδρε, αύριο θα διεξάγουμε μια συζήτηση για την ΑΚΤΑ, ε, για τη συμφωνία αυτή για την καταπολέμηση της παραποίησης. Έχω ένα περιφερειακό κάπως ερώτημα. Μιλάω για τα σχόλια του Επιτρόπου κυρίου Ντεκούχτου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου την 4η 20 Ιουνίου και διαβάζω. Αν αποφασίσετε να καταψηφίσετε ε, την πρόταση αυτή πριν εκδώσει απόφαση το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει ενώπιον του Δικαστηρίου. τέλος της παράθεσης. Νομίζω ότι με τα λόγια αυτά δείχνει ο Επίτροπος ότι δεν γνωρίζει πολύ καλά τις συνθήκες. Πέρα από αυτό, κάτι το οποίο καταγγέλλω είναι το γεγονός ότι εκφράζει μια περιφρόνηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαράδεκτη, μια περιφρόνηση προς τη δημοκρατική διαδικασία και τους πολίτες που εκπροσωπούμε εδώ. Φτάνουμε στο τέλος, λέει η κυρία Πρόεδρος. Νομίζω ότι καταλάβαμε το πνεύμα της ε, παρέμβασής σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάστεξ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο μεγάλο έργο των διδασκάλων, των ε, ε, οικολογικών σχολείων, των, ε, στα πλαίσια του προγράμματος πράσινων σχολείων όπου μαθαίνουν για τις αλλαγές του κλίματος, οι μαθητές μαθαίνουν, σέβονται το περιβάλλον και Πραγματικά με εξέπληξε, με εξέπληξε όταν επισκέφθηκα τα ε, σχολεία αυτά Πόσες πληροφορίες ε, έχουν τα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να επενέσουμε τα σχολεία και το διδακτικό προσωπικό για το έργο τους και θα πρέπει να συστήσουμε στο Κοινοβούλιο να ανταμείψει με βραβείο τους καθηγητές αυτούς που έκαναν τόσο καλή δουλειά σε βάση εθελοντική. Ε, πραγματικά μας ε, περιποιούν τιμή και αξίζουν τον έπαινό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Έμερ Κοστέλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα το χρέος από το τραπεζικό χρέος αποσυνδέθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό και μπορεί έτσι να αποσοβηθεί η κατάρρευση. Όμως ε, δεν ε, ε, πρέπει οι Ιρλανδοί να τιμωρηθούν επειδή ακολούθησαν σόφρονα πολιτική. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε ταχύτερα στις αγορές και αυτό ήθελαν οι Ιρλανδοί όταν στις 31 Μαΐου ψήφισαν τη Συνθήκη Σταθερότητας. Ε, εκείνοι που ε, ε, ψήφισαν όχι, όμως άσκησαν σημαντική πίεση για όλα αυτά. Πιστεύω ότι η Τραπεζική Ένωση, η Φορολογική Ένωση δεν θα πρέπει να παραβλέπει το γεγονός σημασίας ότι είναι πολύ σημαντική η κοινωνική πολιτική. Υπάρχουν ε, πολλά ε, προγράμματα που είναι θετικά όπως τα μέτρα που ε, ενέχουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα ομόλογα έργων κλπ. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο στόχο μιας δικαιότερης κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπή, Θέλω να χαιρετήσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφή τη περασμένη εβδομάδα για τη διάσωση του ευρώ. Να εμφυστήσω την προσοχή σα όμω στα προβλήματα που έχουν οι περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Λουξεμβούργου για να θεωρούνται ως αυτόνομες και ε, έχουσες χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Στη χώρα των Βάσκων εμείς 30 χρόνια τώρα έχουμε στηρίξει την πραγματική οικονομία και έχουμε στοιχηματίσει υπέρ της κοινωνικής οικονομίας, της καινοτομίας ε, και της ε, χρηστής διαχείρισης. Μέχρι πριν από τρία χρόνια ήμασταν ε, οι καλύτεροι στην, στον προϋπολογισμό. Είχαμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και μάλιστα είχαμε και την ηρωνία του υπολείπου ισπανικού κράτους. Και αυτή τη στιγμή υποφέρουμε για κάτι το οποίο δεν αξίζουμε να υποφέρουμε λόγω ενδεχομένως των υπολείπων. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις μέσα ευρωπαϊκά, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή αυτό το οξύμορο και το παράδοξο ε, περιφέρεια ε, με σωστή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση να μην μπορεί να έχει πρόσβαση λόγω των προβλημάτων. Ε, Ο κύριος Χρυσόγελος. σίγουρα εδώ πέρα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρουσε συζητήσει όπω για παράδειγμα για το πολιτέ πρόγραμμα δράση ευρωπαϊκή ένωση στον τομέα τη υγεία για την περιοδο 14 2014-2020 και ένα από του κεντρικού άξονε αυτή τη πολιτική είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών στι υπηρεσίε υγεία. όμω δυστυχώ αυτή την εποχή στην ελλάδα καταραίει το σύστημα υγεία και οι αρχέ τη χώρα έχουν ε, μεγάλε δυσκολίε να διαχειριστούν στοιχειωδώ τι υπηρεσίε υγεία. η κρίση οδήγησε στην αύξηση τη νοσοκομιακή περίθαλψη σε μεγάλο ποσοστό 30% αλλά οι δαπάνε για την υγεία μειώθηκαν κατά 20% ή περισσότερο και καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις και περικοπές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μεγάλο κομμάτι των πολιτών μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εξαιτίας ανεργίας και των περιοριστικών πολιτικών μένει εκτός του συστήματος υγείας. το προεδρείο της ομάδας των πράσινων παρέδωσε πρόσφατα επιστολή στον κύριο μπαρόζο για να λάβει δράση και να διασφαλίσει ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ζωής των πολιτών κάθε άνθρωπος στην ελλάδα θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια και να έχει πρόσβαση σε ποιοτική ε, προληπτική περίθαλψη και δικαίωμα σε ιατρική θεραπεία και νομίζουμε ότι η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να επανεξετάσει όρου του μνημονίου έτσι ώστε να γίνει συμβατέ με τι ευρωπαϊκέ αξίε και πολιτικέ. Ευχαριστώ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Δούμα ασχολείται με τις χώρες που την περιβάλλουν. Ασχολήθηκε με την ε, Λετωνία και τη Λιθουανία. Οργανώθηκαν επίσημες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Ρωσία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία. Πριν από μερικές μέρες η Ουγγρική η Κοινοβουλευτική Επιτροπή οργάνωσε με προκλητικό τρόπο μία συνάντηση στη Σλοβακική, στο σλοβακικό έδαφος. Τους ε, δόθηκαν χωρίς προειδοποίηση αίθουσες του Πανεπιστημίου και συζητήθηκε το θέμα των Ούγγρων που ζουν στη Σλοβακία. Δεν θα ήταν ε, σκόπιμο για το διπλωματικό πρωτόκολλο να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχουμε 26 ανεξάρτητα κράτη και μία απικία. Την αγαπημένη μου πατρίδα, την Ρουμανία, που είναι αμερικανική, όπου οι πράκτορες της υπαδρούν ε, δρούν ως δουλέμποροι και έχουν τρεις ε, βασικούς στόχους. Να λαιλατίσουν τον πλούτο της χώρας, χρυσό, άργυρο, ουράνιο και φυσικό αέριο της χώρας. Δεύτερον, να αναγκάσουν τους Ρουμάνους να τους αναγκάσουν να αγοράσουν 46 F-16 του από το 65 και τέλος μια ειρηνική χώρα τη Ρουμανία να την βάλουν να παίξει το ρόλο της αντιπυραυλικής ε, ασπίδας ενάντια στη Ρωσία. Η τελευταία ε, απάτη έγινε στις τελευταίες τοπικές εκλογές όπου πάνω από 90 στελέχη της CIA ε, ήταν αναμεμειγμένα στην, ε, στο στήσιμο των εκλογών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα κάθε κράτος μέλος της αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές. Η, αυτή τη στιγμή είναι ζωτική σημασία να συνεργαστούν σωστά και στενά τα κράτη-μέλη, να έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις σε αμοιβαία βάση. Οι εταιρικές σχέσεις οι συνεργασίες θα πρέπει να είναι το, πιστεύω, το βασικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και ανησυχώ ιδιαιτέρως διότι το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ε, λειτουργήσε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε σε επικράτεια που εντάσσεται στην εθνική κυριαρχία της Σλοβακίας. Αυτό είναι κατακριτέο. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβακίας κάνει το παν για να καλλιεργήσει τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και θα πρέπει η Ουγγρική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι πήγα στη Washington και συνάντησα εκπροσώπους και των δύο κομμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όπως γνωρίζετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ψήφισαν για να υποστηρίξουν αυτό τον νόμο και εδώ στην Επιτροπή Ξένων ε, Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσουμε την έκθεση Μαγνίξη. Η πρόταση είναι παρεμφερής με αυτό που εξετάζεται τώρα στις ε, Μεγάλη Βρετανία σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά εγκληματικές ε, οργανώσεις από τη στιγμή που τα άτομα αυτά κινούνται ελεύθερα στην Ευρώπη αλλά πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Διαμαρτύρομαι κατά των καταχρήσεων ε, στη Ρουμανία από τους κρατικούς φορείς ε, και τη δικαστική εξουσία και τις μυστικές υπηρεσίες. Ε, ο πρόεδρος και η πρώην δεξιά διακυβέρνηση χρησιμοποίησε τους φορείς αυτούς για, ως μέσον ελέγχου κατά αυτής της κυβέρνησης. Ε, ο σκοπός είναι να παρεμποδιστεί το έργο της παρούσας κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο ε, απέκλεισε τον Πρωθυπουργό από την άσκηση των προνομίων του. Βλέπουμε ε, παρενόχληση ε, γιατρών αστυνομικών επειδή κάνουν τη δουλειά τους έτσι υπονομεύουν το κράτος δικαίου και αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια εκστρατεία από, τα, από τους θεσμούς ε, παρά το Προέδρο και το ΕΛΚ τους υποστηρίζει. Ε, Ευχαριστώ κυρία Ντανσίλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη Ρουμανία έγινε πραγματικά μία αλλαγή μετά τις εκλογές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια, να δούμε γιατί έγιναν οι παρεκκλήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, να προτείνουμε ένα νέο μοντέλο και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την καταψήφιση της πρότασης των μελών του Κοινοβουλίου του PDL. Αυτή τη στιγμή παγιώνεται η δημοκρατία στη Ρουμανία. Και ο ρουμανικός λαός αυτή τη στιγμή κάνει βήματα προς τα εμπρός. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας επίσης διότι το Ρουμανικό Κοινοβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να συζητήσει τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια αλλαγή αυτή συγκριτικά με τη στάση του προκατόχου του προηγούμενου Προέδρου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλεχερ έχει το λόγο. Χαιρετίζω την ε, έκβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, είναι πολύ σημαντικός ο νέος ρόλος ε, για τις τράπεζες. Η συμφωνία είναι σημαντική για την Ιρλανδία και την αναδιάρθρωση του χρέους που θα οδηγήσει σε μείωση του ε, βάρους στους φορολογουμένους. Καταλαβαίνω ότι οι Υπουργοί Οικονομικών θα κάνουν διαπραγματεύσεις και σχετικά με το χρέος της Ιρλανδίας. Ε, και θα υπάρξει ισορροπία απέναντι στην Ισπανία, Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα του δημοψηφίσματος για την πρόσβαση στον ESM. Ε ε, είναι πολύ σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για την Ιρλανδία και την Ευρωζώνη, ο ESM και ε, η αποσύνδεση του τραπεζικού από το δημόσιο χρέος είναι πολύ σημαντικό για τα βήματα μπροστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις εβδομάδες Πρόκειται να γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ με στις, ε, στην τελευταία συνάντηση, στη συνάντηση του Βουκουρέστι με προσώπους με των Ρουμάνων Γεωργών, τονίσαμε τις προσδοκίες που υπήρχαν ως προς την πρόταση της Επιτροπής μαζί με τους σοσιαλιστές συναδέλφους. Θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι οι αποφάσεις αυτές θα λάβουν υπόψη τους τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ιδιαίτερα αναπτυγμένων γεωργιών ορισμένων σχολών μπελών και άλλων λιγότερο ανεπτυγμένων ε, γεωργιών. Ε, επικροτώ την έκθεση του κυρίου κάπου Σάντος που ζητάει μια πιο δίκαιη κατανομή των άμεσων πληρωμών έτσι ώστε οι χώρες μέλη που έχουν χαμηλότερες πληρωμές να μπορέσουν να ε, ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. παρακαλούμε. Μετά από 7 χρόνια ταμείου ανεργίας η... στην ε, Ανάνη, μία από τις βασικές εταιρείες, κηρύξε πτώχευση και ξεκίνησαν ε, απολύσεις 1.300 ατόμων. Ε, η δεύτερη μεγάλη επιχείρηση της περιοχής ε, Λάτσιο κλείνει και ε, πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία αγοράστηκε με στόχο να οδηγηθεί σε πτώχευση και να μεταφερθεί η παραγωγή σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον για αυτές τι επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι διανύουν μία περίοδο κρίσης. Εδώ και 7 χρόνια αντιμετωπίζουν ανασφάλεια στην ε, ε, επαγγελματικά. Θα πρέπει να θέσουμε σε φαρμαγή όλα τα απαραίτητα μέσα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε εργασία και παραγωγικό μέλλον σε αυτό το σημαντικό συγκρότημα. Ευχαριστώ κύριε Άντζερ, ο κύριος Κόρκας Λάστρα. Θα ήθελα να καταγγείλω το όραμα που έχει η Ισπανική κυβέρνηση για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μην γίνουν περικοπές στον κλάδο της έρευνας και της καινοτομίας. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση έκανε περικοπές 22%. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερους ερευνητές, να σταματήσουμε τη διαρροή εγκεφάλων προς το εξωτερικό για να μπορέσει η χώρα να ανακάμψει. Είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται μόνο ελάχιστοι και να περικόπτεται ο αριθμός των υποτροφιών. 1,2 του ΑΕΠ ε, αφιερώνουμε μόνο στην έρευνα. Ε, με αυτή την έννοια δεν είναι δυνατό να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο. Η Ισπανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επιμένει ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμό του επιστημονικού προσωπικού, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι το βασικό κεφάλαιο για την ανάκαμψη τη οικονομία. Επιμένω λοιπόν οι επιστήμες, η τεχνολογία θα πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και να μην έχουμε την κρίση ως δικαιολογία για να κάνουμε περικοπές. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση λόγω της απελευθέρωσης των, του Εστέμπαν Περάλτα Λοσίγια μαζί και με άλλα τρία άλλα μέλη της αντιπροσωπείας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου. Αυτοί οι νομικοί σύμβουλοι έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και υπάρχει βεβαίως και το αρνητικό νέο, το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιλότους των ελικοπτέρων ε, οι οποίοι μάχονται για την κατάσβεση των ε, πυρκαγιών, των πυρκαγιών στη Βαλένθια. Έχουμε έλλειψη στις επενδύσεις, στις επενδύσεις στο κράτος, στις δημόσιες υπηρεσίες, εξού και οι πυρκαγιές στην Ισπανία ε, φέτος ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απελευθέρωση του Εστέμπαν Περάλτα και να εκφράσω τη λύπη μου για τον θάνατο του άτυχου πιλότου ελικοπτέρου. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει ο κύριος Κουσκιέρη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για το πρόβλημα της ε, ε, λάθρο στη Μάλτα να σας πω ότι έχει οξυνθεί τα τελευταία ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Πολλοί αφήνουν τις χώρες τους στην Αφρική προσπαθώντας να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη και έχουμε ε, ε, αύξηση των ανθρώπων που έχουν μπει στη Μάλτα παρανόμως. Θέλω να σας καλέσω να επιδείξετε μεγαλύτερη λυλεγγύη στη Μάλτα είναι μια πρόκληση για όλη την Ευρώπη και δεν θα πρέπει το βάρος αυτό να το φέρει μια μικρή νησιωτική χώρα η Μάλτα που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στις δύο Υπήρους. Δεν μπορούμε να το ε, αναλάβουμε μόνοι μας αυτό το βάρος και η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποτύχει, δεν λειτουργεί. Πολύ λίγα κράτη-μέλη προσφέρουν τη βοήθειά τους σε εμάς στη Μάλτα. Ενώ υποχρεούνται τα κράτη-μέλη εξ ονόματος της αλληλεγγύης να κάνουν ένα βήμα προς το εμπρός. Χρειαζόμαστε αυστηρούς κανόνες που να εφαρμόζονται από όλους και παντού. Άλλωστε η Μάλτα συμβάλλει και συνεισφέρει στο μηχανισμό αυτό. Θα πρέπει να μοιράζονται τα βάρη και να είναι αποτελεσματικός αυτός ο μηχανισμός. Ευχαριστώ. Θα εξετάσουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Πόλσεν για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων από το